Καλή σας μέρα. Μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Και όμως, δεδομένης της απόφασης που πήραμε στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην ένταξη του επόμενου σημείου στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα φάρμακα ε, χωρίς ε, πατέντα στα πλαίσια της μελλοντικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Επίσης, η ακρόασή μας για αύριο είναι εκπαίδευση για την ανάπτυξη και όχι εκπαίδευση και ανάπτυξη. Έχετε σχόλια για την τροποποίηση αυτή στην ημερήσια διάταξη μήπως? Όχι, εγκρίνεται συνεπώς η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 12 η και 13 η Ιουλίου 2011. Τα έχετε όλοι στη διάθεσή σας. Αν έχετε παρατηρήσεις επί των πρακτικών αυτών, παρακαλώ να ενημερώσετε τη γραμματεία πριν από τη λήξη της σημερινής μας συνεδριάσεως. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ερωτήσεις δεν έχουν υποβληθεί για να υποβάλουμε και εμείς με τη σειρά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ όμως έχω μία ανακοίνωση να κάνω στο σημείο 4, στις ανακοινώσεις δηλαδή της Πρόεδρου δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας χωρίς να αναφερθούμε στην Λιβύη και στο δράμα που περνάει το κέρδος Αφρικής. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Διάφορες υποδομές έχουν καταστραφεί στη Λιβύη, ιδιαίτερα όσον αφορά το νερό και τον ηλεκτρισμό. Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις αιστείες τους και βρίσκονται στα σύνορα με γειτονικέ χώρες, όπως για παράδειγμα στα σύνορα με την Τινησία. Από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά θύματα μετά από μάχες, οι οποίοι μπορεί να έτυχε να βρέθηκαν την κακή στιγμή στο κακό σημείο. Πρέπει να υπάρξουν έργα ανοικοδόμησης όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα έργα αυτά είναι τεράστια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει τον ρόλο που της πρέπει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε να έρθει και να μας ε, ενημερώσει για το ποια είναι τα έργα που προβλέπει να αναλάβει και τι μέσα θα κινητοποιήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την κρίση αυτή. Έρχομαι τώρα στην περίπτωση του κέρατος της Αφρικής. Η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Εδώ και μισό αιώνα ο κόσμος υποφέρει από λοιμό. 12 εκατομμύρια άνθρωποι ε, βρίσκονται σε κατάσταση να μην έχουν αρκετά τρόφιμα, ζουν σε καταβλισμούς προσφύγων, ε, όπου βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος, ε, πιεσμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Και εδώ θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθούν λύσεις με τα 27,5 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν επιπλέον από αυτά που ήδη έχουν αποφασιστεί φέτος. Πρέπει να ετοιμαστεί ένα νέο σχέδιο με 60 εκατομμύρια ευρώ και η αποστολή που έχει αναλάβει επιτόπου η κυρία Ζωζιέβη είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε γιατί. Υπάρχει, ε, γιατί έχουμε οδηγηθεί εκεί, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη ξηρασία, γιατί αυξάνονται οι τιμές των φυσικών πόρων. Δεν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί μια τέτοια καταστροφή. Ίσως τα μηνύματα που είχαμε από πριν ε, να έπρεπε να τα έχουμε πάρει πιο σοβαρά υπόψη μας και να μπορούσαμε έτσι να είχαμε αποφύγει αυτή την κατάσταση και μια κερδοσκοπία η οποία μαστίζει την περιοχή και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ήρθε η στιγμή όντως να ανασκουμποθούμε και να φροντίσουμε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ίσως πρέπει να δημιουργηθεί μια παγκόσμια υπηρεσία για τη ρύθμιση των αγορών και για αποθέματα σιτηρών και άλλων τροφίμων, κάτι το οποίο προτείνει ο ειδικό εισηγητή του ΟΕΕ και έχουμε και εμεί εγκρίνει. Όπω επίση και μηχανισμού αλληλεγγύη που να μπορούμε να εφαρμόσουμε εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιε λύσει πρέπει να καθίσουμε να τι σκεφτούμε. Είναι ήδη ένα μέρο τη δουλειά που έχει ήδη κάνει η Επιτροπή μα και θα συνεχίσει να κάνει, ιδιαίτερα με την ακρόση τη 4η Οκτωβρίου που έχει να κάνει με την επισητιστική ασφάλεια. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει εμένα όλου ιδιαίτερω. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα με τη σειρά της ανακοινώσει να μας κάνει. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Κατερίνα Ματεβάντικεν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κατερίνα Ματεβάντικεν, ονομάζομαι όντω, ονομάζομαι, ε, δουλεύω στην ε, Γενική Διεύθυνση ΑΦΚΟ και έχω αναλάβει τον ε, διοργανικό συντονισμό. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα αυτή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω είναι ανακοινώσω τα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη. Έχουμε τρεις ανακοινώσεις που θα υιοθετήσουμε κατά τα τέλη του Οκτωβρίου. Η πρώτη ανακοίνωση, πιο σημαντική, είναι ανακοίνωση για την ε, πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δημόσαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από πέρυσι, ε, βάσει πράσινης βίβλου, ξεκίνησε διαβούλευση με το κοινό όπου συμμετέχουν εταίροι από ολόκληρο τον κόσμο για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή μας ε, στη συνεργασία και την ανάπτυξη. Ε, προσπαθούμε να πάρουμε μαθήματα και από τη διαβούλευση αυτή αλλά και από την Αραβική Άνοιξη βέβαια. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, μόνο θα σας μεταφέρω κάποιες ιδέες που φυσικά και θα μας βοηθήσουν να υιοθετήσουμε στρατηγική, τη στρατηγική μας. Η Επιτροπή θέλει να επικεντρώσει τη βοηθειά της στοχευμένα ε, σε διάφορες χώρες Θέλουμε επίσης να επικεντρωθούμε περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα και προτείνουμε και μη διαφοροποιημένη προσέγγιση. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε κοινέ στρατηγικές Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατημέλη και να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα και το εύρος τους ενισχύοντας την διαφάνεια στην ε, συνεργασία. Υπάρχουν και δύο άλλες ανακοινώσεις που ετοιμάζουμε. Πρόκειται για μια κοινή θέση για την Βουτσουάνα πρώτον, πώς να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της αρρωγής μας. Πώς θα εφαρμόσουμε τις αρχές μας, τους διάφορους παράγοντες και πώς θα υποφεληθούμε ακόμα περισσότερο από την χρηματική οικονομική ενίσχυση. Τέλος, ετοιμάζουμε και τελειοποιούμε τώρα μία ανακοίνωση για την δημοσιονομική στήριξη. Πώς δηλαδή θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές από τη συνθήκη της Λισαβόνας και πώς το μέσο αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται στην εμπειρία που έχουμε και από τα αποτελέσματα που έχουμε από την δημόσια διαβούλευση. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται βάσει ανακοίνωσης του Ιουνίου του 2011 για τις δημοσιονομικές προοπτικές όσον αφορά την περίοδο 2014-2020. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω στα διάφορα αναπτυξιακά μέσα και θα επανέλθουμε εδώ με περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα τις έχουμε τα κύρια στοιχεία για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές όσον αφορά την ανάπτυξη είναι πρώτα απ' όλα το όριο του 0,7% του ΑΕΠ που θέλουμε να διατηρηθεί ως ε, ποσοστό για την αναπτυξιακή βοήθεια των ε, χωρών μελών. Κάτι άλλο σημαντικό είναι το 15 εκτός προπολογισμού για αυτή την περίοδο. Και τελειώνω με μια μικρή ανακοίνωση. Ότι δηλαδή ετοιμάζουμε τις σημερίδες ε, αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβουν χώρα το Δεκέμβριο στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Τώρα περνάμε στα σημεία 6 και 7 που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την βιομάζα και αντίκτυπός της στην ανάπτυξη. Πρόκειται για ερώτηση που ζητάει προφορική απάντηση και πρόταση ψηφίσματος. Τον Απρίλιο του 2009 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε οδηγία η οποία καθορίζει κοινό κοινοτικό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας που προέρχεται από εναλλακτικέ ε, πηγέ ενέργεια. Πρόκειται για την οδηγία 28 του 2009. Στόχο είναι το 2020 να πετύχουμε 20% ενέργεια από ανανόσιμες πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 10% ενέργεια από ανανόσιμες πηγές ε, ενέργειας σε κάθε κράτος μέλος. Και ενώ υπάρχει όλο και μεγαλύτερη παραγωγή και χρήση της βιομάσας, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κανένα σταθερό πλαίσιο το οποίο να διασφαλίζει την παραγωγή και την βιώσιμη χρήση της βιομάσας για την ενέργεια. Έπειτα, μερικές φορές η βιομάζα που προέρχεται από ξύλο έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφονται δάση για να γίνονται ενέργεια και βιοκαύσιμα. Στόχο λοιπόν της προφορικής αυτής ερώτησης και του ψηφίσματο είναι να ξεκινήσει η συζήτηση για να δούμε τι μέτρα σκοπεύει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η βιομάζα που χρησιμοποιείται για την ενέργεια είναι βιώσιμη και συμβιβάζεται με μια επίσης καλή αντιμετώπιση των δασών για να μην καταστρέφονται αυτά. Θα σας δώσω το λόγο σε όλους για αυτό το θέμα. Πάντω να ξέρετε ότι είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη, γι' αυτό και θα σας περιορίσω δύο λεπτά ο καθένα για ό,τι παρατηρήσεις έχετε. Η κυρία Όιλ πρώτα, για δύο λεπτά παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, χαιρετίζω αυτή την ε, προφορική ερώτηση και πιστεύω ότι έχουμε δίκιο που την θέτουμε και που ζητούμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω απλώς είναι να προτείνω ορισμένα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αν είναι δυνατόν να την τροποποιήσουμε και ζητούμε μία σημαντική αύξηση στη χρήση της βιομάζας Τώρα όμως έχουμε <clears throat> το πρόγραμμα δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό να έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούνιο. Οπότε ε, είναι δυνατόν να δούμε τι πρόκειται να κάνουν οι χώρες και ε, ποια είναι τα προγράμματα τα οποία διατυπώνουν που πρέπει να διπλασιάσουν τον τομέα αυτό μέχρι το 2020. Θα πρότεινα λοιπόν να περιληφθεί στο κείμενο γιατί θα έχουμε έτσι μία ιδέα για την κλίμακα μεγέθους του προγράμματος. Επίσης θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να προβεί σε μία αναθεώρηση. Μία αναθεώρηση σχετικά με ε, τα ε, κριτήρια αηφορίας για την βιομάζα και τα βιοαέρια μέχρι το τέλος του 2011 και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά. Ζητούμε όμως να λάβουν υπόψη επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της ε, συνεκτικότητας με την βιοπικιλότητα και με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στον τομέα αυτό κατά τρόπον ώστε η Επιτροπή μέσα σε αυτή την αναθεώρηση να περιλάβει και τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκρέσ. Ε, ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω πολύ γρήγορα ότι χαίρομαι πολύ με τη λύση η οποία έχει προταθεί από τη Γραμματεία. Καταρχήν τονίζει ότι δεν υπάρχει ένα ισχυρό πλαίσιο και πρέπει να συνδυάσουμε τα, τα κριτήρια σχετικά με τη βιομάζα. Ε, επίσης ε, δεν έχει ληφθεί υπόψη ε, την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλάβει μία μεθοδολογία κατά τρόπον ώστε θα μπορούμε μπορέσουμε να περιλάβουμε τα κριτήρια υπολογισμού της ε, καταναλώσεως και ε, να λάβουμε υπόψη την κατανάλωση και την αποτελεσματικότητα ε, της ενεργείας και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ καλά θέματα που αναφέρονται στο ψήφισμα της βιομάζας. Ευχαριστώ. Το, ημερομηνία Μάλλον με συγχωρείτε, ε, ε, πρέπει πρώτα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Hans Van Senden. Ευχαριστώ. Ε, χαίρομαι που θέσατε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη διότι είναι ένα θέμα το οποίο χαίρει της πλήρους προσοχής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ορισμένα από τα θέματα τα οποία αναφέρατε στο ερώτημά σας ε, πρέπει ίσως να επεκταθούν. Θα ήθελα να ξέρω, θέλετε να ε, απαντήσουμε τώρα, σκοπεύετε Θέλετε να απαντήσετε αμέσως. Δεν έχουν γυρίσει όλοι οι υπεύθυνοί μας επί του θέματος από τις διακοπές, οπότε περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Euh, λοιπόν, καθορίσαμε μία ημερομηνία για την υιοθέτηση του κειμένου και ε, του ψηφίσματος οι τροπολογίες ε, στις 5 Σεπτεμβρίου και ε, η ψήφιση του κειμένου θα είναι για τις 22 Σεπτεμβρίου. Τώρα, επόμενο θέμα, τα, η φραγμή στις ανταλλαγές και στις, α, επενδύσεις. Ε, ε, το λόγο έχει η κυρία Σαρκεντίνη, ε, η οποία θα παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως αυτό το οποίο έχετε εδώ είναι μία γνωμοδότηση ε, της Επιτροπής μας στην Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με τις διάφορες εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 που βασίζονται στην ε, προηγούμενη πρότασή τους σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις. Η πράσινη έχουν ε, διατυπώσει αυτή τη γνωμοδότηση, τη σύντομη γνωμοδότηση και θα ήθελα να σας πω ότι ευχαρίστω θα ακούσω μέχρι τις 31 Αυγούστου 12 το μεσημέρι ε, τις τροπολογίες σας ε, πέστε ό,τι χρειάζεστε διότι είναι πολύ σύντομη για να μας τα πει όλα ε, και εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένες τροπολογίες στην έκθεσή μου και αυτό που προσπαθώ να τονίσω είναι αυτό που προσπαθούμε πάντοτε να τονίσουμε όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και την ανάπτυξη, δηλαδή τη συνεκτικότητα της ε, ε, αναπτύξεως. Ε, υπάρχει ένα άρθρο της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, που τονίζει ότι δεν πρέπει ε, να, να εμποδίζουμε την επίτευξη του βασικού μας στόχου που είναι η μείωση της φτώχειας και η ανάπτυξη. Και η Επιτροπή μας ε, αναφέρεται σε ορισμένα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ινδία, πρώτων υλών στην Κίνα και προσπαθώ να τα περιλάβω στη γνωμοδότηση αυτή λέγοντας ότι οι υποανάπτυξη χώρες και οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τις αγορές τους. Αυτό το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ελεύθερο εμπόριο θα είναι προς όφελος όλων μας μου υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε μία ελεύθερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε ευτυχείς που δεν έχουμε ε, ελεύθερη αγορά και ε, προσπαθούμε να να πιέσουμε τις άλλες χώρες να προβούν σε μία απελευθέρωση της αγοράς. Πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ε, τις ε, ε, τις επιλογές τους να μπορούν να επέμβουν εις τις διαπραγματεύσεις του ΓΚΑΤΣ και ε, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητάμε για πρώτη φορά σχετικά με την επιρροή του εμπορίου στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόλ έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζω την προσπάθεια αυτή και όντως θέλω να κάνω μόνο ένα σχόλιο. Νομίζω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα στην παράγραφο 3 είναι η πίεση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για να ε, ε, αποβάλουν τους την εξαγωγική φορολογία και ε, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός καταλόγου αναπτυσσομένων χωρών και της Κίνας. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μία επιπλέον παράγραφος επί του θέματος διότι η Κίνα η οποία θέτει φραγμούς στο εμπόριο είναι τρομερό. Το πράττουν για να προστατεύσουν την εσωτερική τους και καταρτίζουν πολύ ε, σοβαρά ε, εμπόδια ε, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ανανεώσιμα ε, προϊόντα όπως είναι παραδείγματο χάρη τα ηλιακά κάτοπτρα να υφίστανται μεγάλη φορολογία και ε, ε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην υποστούν αρνητικές επιπτώσεις οι εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία τροπολογία και να συμπληρώσω το θέμα αυτό ε, σχετικά με το θέμα ε, των φραγμών των υποανάπτυξη χωρών οι οποίες ναι μεν χρειάζεται να προστατεύουν τις αγορές τους αλλά χωρίς υπερβολές. Ο κύριος Γκέρνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν για τις συμφωνίες ε, της οικονομικής εταιρικής σχέσης ιδιαίτερα με τις χώρες ΑΚΕ. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Τι κάνετε στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. Μια χώρα που δεν έχει μεγάλα φορολογικά έσοδα φέρει πίν σκοπεύετε να έχετε μια ειδική μεταχείριση για τη χώρα αυτή δίνοντα την ιδιότητα να έχουν παραδείγματο χάρη πιο ψηλού δασμού για να εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Γιατί είναι χώρε οι οποίε δεν έχουν καθόλου λεφτά και χρειάζονται αυτά τα έσοδα για να λειτουργήσει ο προπολογισμό του. Δεύτερον, τα ΑΠΤΙΚ. Κατά την άποψή σα ή από ό,τι ξέρετε, υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, ιδιαίτερα στα φάρμακα ρετροβίρους, επειδή δεν εφαρμόζεται πλήρως η συμφωνία BDIC. Γνωρίζετε αν υπάρχουν χώρες οι οποίες στερούνται αυτής της δυνατότητας λόγω των διατάξεων όσον αφορά την εφοδιασμό τους σε φάρμακα που είναι απολύτως αναγκαία για την καταπολέμηση τόσο σοβαρών ασθενειών. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ποιος θέλει να απαντήσει. Μάρτιν Μπίσοφ λέγομαι από τη Γενική διάθεση για το Εμπόριο. Μονάδα πρόσβαση στην αγορά. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας δώσετε τη δυνατότητα να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε την γνωμοδότησή σας. Η έκθεση αυτή για τους φραγμούς, εμπορικούς κλπ. δεν έχει στόχο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αναφέρεται κυρίως στους πιο σημαντικούς εταίρους μας, εμπορικούς εννοώ εταίρους. Και η έκθεση δείχνει τη σχέση μας με τις χώρες αυτές πως οι διεθνείς υποχρεώσεις και δικαιώματα φυσικά και των δύο πλευρών τηρούνται ή όχι στις διεθνείς συμφωνίες γιατί διακυβεύονται πολύ σημαντικά οικονομικά ποσά. Θέλουμε να υπάρχει αξιοπιστία στην ημερήσια διάταξη εφαρμογής των μέτρων αυτών εκ μέρους μας Θέλουμε να το συντονίζουμε με τα κράτη-μέλη, αυτό είναι η πολιτική ημερήσια διάταξη, να αρθούν οι εμπορικοί, τα εμπορικά εμπόδια που δεν θα έπρεπε καταρχήν να υπάρχουν καν. Μπορώ να σας πω το εξή. Πρώτον, όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξη. Αυτή είναι η εμπορική πολιτική για την πρόσβαση στις αγορές. Συντονιζόμαστε με την πολιτική ανάπτυξη της Κομισιόν. Η δική μας στρατηγική, επαναλαμβάνω, δεν έχει σε στόχο τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Καθόλου. Η έκθεση καλύπτει τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις αναδυόμενες οικονομικά χώρες που έχουν ήδη θέση διεθνώς και είναι μέλη του ε, Παγκόσμιου Οργάνωση Εμπορίου. Στόχος, όπως ξέρετε, είναι να, είναι να δίκαιο εμπόριο και για τις δύο πλευρές. Όσο πιο ασθενής λοιπόν είναι μια χώρα, τόσο πιο σκόπιμο είναι να έχει μια καλή θέση μέσα στο πλαίσιο αυτό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πιο μικρές χώρες, όπου το περιβάλλον είναι πολύ καλύτερο παρά να μην υπήρχαν κανόνου κανόνες. Στην ερώτηση σχετικά σχετικά με την ε, Ινδία, την Κίνα κλπ. Η Ινδία και η Κίνα λόγω των υποχρεώσεων τους με βάση τις διεθνείς συνθήκες και αυτό εξάλλου αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Η έκθεση δεν είναι η εφαρμοζόμενη πολιτική, απλώς περιγράφει το τι γίνεται στην πραγματικότητα και κατά πόσον η Κομισιόν μπορεί ή όχι να παρέμβει σε συντονισμό πάντα σε μια πολιτική ε, που συμφωνεί με τις άλλες πολιτικές της Κομισιόν και κυρίως με την πολιτική ανάπτυξης. Για την ερώτηση σχετικά με την πίεση της ε, ε, εξαγωγικούς φόρους και λιγότερα αναπτυγμένες χώρες. Οι χώρες αυτές με βάση την πολιτική ανάπτυξη και τις προτεραιότητες λαμβάνονται διόντως υπόψη και στις επιμέρους συμφωνίες της στις διαπραγματεύσεις μας απόλυτα με την πολιτική ανάπτυξη με οτιδήποτε δυνατότητα ευελιξίας αυτό μας επιτρέπει ως προς τους εταίρους μας αυτούς. Για τις διαπραγματεύσεις είπα αν έχουμε ίση μεταχείριση ή αν μια χώρα μπορεί να αυξήσει τους δασμούς. Ειδικά οι διαπραγματεύσει αυτές, είπα, δείχνει το πόσο συζήτηση γίνεται μεταξύ της Κομισιόν και τις συγκεκριμένες αυτές χώρες και περιφέρειες στην οποία ανήκουν. Επαναλαμβάνω όλα τα μέτρα ε, ευελιξίας λαμβάνονται υπόψη. Το ίδιο και τη συμφωνία τρίψη. Συγγνώμη, αλλά από ό,τι ξέρω, καμία χώρα δεν έχει απαγόρευση πρόσβαση στα φάρμακα λόγω της εφαρμογής της συμφωνίας TRIPS. Ευχαριστώ. Είναι δυνατόν η Κομισιόν να μας δώσει πληροφορίες, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Πάμε χάρη για την εφαρμογή της συμφωνίας TRIPS. Γιατί ακούμε διεστάμενα μηνύματα ανάλογα από πού έρχεται το μήνυμα. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή θεσμικούς φορείς. Δεύτερον, για την ευελιξία Συμφωνώ, μάλλον ε, δέχομαι αυτό που είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν σχετικά με την ευελιξία που επιδεικνύει στι διαπραγματεύσει της Κομισιόν. Όμω, λειτουργείται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι φορεί που να ασκήσουν πίεση στο επίπεδο φορολόγηση φερειπίν των συγκεκριμένων χωρών. Παραδείγματο χάρη το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή η Παγκόσμια Τράπεζα μπορούν και αυτοί να βάλουν όρους που κατά να μην συγκλίνουν με την άποψη της Κομισιόν. Και εδώ θα ήταν χρήσιμο εμείς ως πολιτικοί που είμαστε να ξέρουμε ποια είναι η άποψη των άλλων αυτών φορέων που δεν συμφωνούν με την Κομισιόν. Από ό,τι θυμάμαι, θυμάμαι ένα επεισόδιο με θύμα την Γκάνα πριν από 8 χρόνια ήθελε να εφαρμόσει πιο ψηλούς δασμούς και νομίζω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την έπιασε όμοιρο κυριολεκτικά τη χώρα αυτή με ένα δάνειο που είπε θα σου δώσω το δάνειο Μεξικό αν μειώσει τη φορολόγηση αυτή. Αν λοιπόν άλλοι πέραν της Κομισιόν μπορούν να παρεύουν όσον αφορά την ευελιξία δράσης που αναφέρατε, χρήσιμο είναι να το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Χολ. Έφυγε, αλλά συμφωνώ με αυτό που είπε. Φυσικά συμφωνώ να γίνει η διαφορά μεταξύ λιγότερα αναπτυγμένες χώρε και αναδυόμενε χώρε. Το είπε και η Κομισιόν. Ξέρω ότι η Κομισιόν ε, εδώ ε, σημειώνει ιδιαίτερα ορισμένε αναδυόμενε χώρε. Όσον αφορά όμω το εμπόριο και την επενδύσει, κλπ. Καλό θα είναι να προειδοποιήσουμε το πώς θέλουμε να γίνεται, να εξελίσσονται οι σχέσει μας με τις λιγότερα αναπτυσμένες χώρε. Η Ινδία ως αναδυόμενη χώρα. Ναι, αλλά έχουμε δυσκολίες. Φάρμακα, παραδείγματος χάρη, της Ινδίας δεν βρίσκουν αγορές στο εξωτερικό λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ. Μια άλλη απάντηση προς την Κομισιόν. Αν όλες οι χώρες αυτές είναι μέρος του ΠΟΗ, που είναι, Ποιο ο λόγος να πιέζονται να έχουν διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές και να μην μένουμε στις διεθνείς συμφωνίες. Και τελειώνουμε το εξή. Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη μη ανακόλουθες πολιτικές εννοούμε μία ανακόλουθες όσον αφορά την ανάπτυξη. Χαίρομαι για το ότι η Κομισιόν έχει μία εσωτερική πολιτική, μία ανακόλουθη όσον αφορά το εμπόρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μία ανακόλουθη για την ανάπτυξη. Αφορά εσά το εσωτερικό της λειτουργίας σας που δεν είναι το ίδιο. Εγώ αναφέρομαι να υπάρχει μία ανακολουθία όσον αφορά την ανάπτυξη. Για τις τροπολογίες σε δύο μέρες, στις 12 η ώρα, λίγη προθεσμία. Και, αν έχετε, και Όλα τα σχόλιά σα, ήταν πάρα πολύ εύστοχα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, τονίζω και εγώ αυτό που είπε η κυρία Σαργεντίνη. Κατάθεση τροπολογιών 31 Αυγούστου 12 η ώρα. Ψηφοφορία στι 22 Σεπτεμβρίου. Τώρα φτάνουμε στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης. Στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και ξεπερνώντας τις δυσκολίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση της Επιτροπής ΑΦΕΤ, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, είναι αρκετά ισορροπημένη και πλήρης. Εγώ σας προτείνω μια γνωμοδότηση που ζητάμε να λάβει υπόψη της Επιτροπή ΑΦΕΤ και σε αυτήν σημειώνω ορισμένα σημεία ε, τα οποία θα θέλαμε να τονίζονται περισσότερο στην τελική έκθεση, γιατί είναι υψηλή δικιά μας πολιτική προτεραιότητα. Βέβαια το κείμενό μας δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό προφορικά θα προσθέσω ορισμένα πράγματα σε αυτά που έχω ήδη βάλει γραπτά. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να χρησιμοποιούν ό,τι διπλωματικά μέσα έχουν στη διάθεσή τους για να προωθούν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να το προωθούν στις ε, διάφορες χώρες και να επιμείνουν σε αυτές που δεν το έχουν ακόμα, που δεν έχουν κυρώσει την ιδρυτική του πράξη, να το κάνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι ε, προς όφελό μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε ε, τις άλλες χώρες και κυρίως τις χώρες εκεί για τη σημασία που έχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έπειτα είναι πολύ βασικό να υπάρχει μια συνοχή στην εξωτερική μας πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί τη δημοκρατία, μια δικαιοσύνη αμερόληπτη και ανεξάρτητη και να προωθεί επίσης και να υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τίποτα δεν πρέπει να την εμποδίζει από το στόχο αυτό, ούτε καν τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, όπω είδαμε στην Τινησία ή στη Λιβύη. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε ηγέτε οι οποίοι καταπιέζουν το λαό του με σκοπό να αυξάνουμε το ευρωπαϊκό ΕΠ. Στη συνέχεια θα ήθελα ρητά να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από όλες τις χώρες ε, μέλη της συμβαλόμενας της διοικητής ε, Κοπεχάγης, τη Γενική Εισαγγελία κλπ. να ενισχύσουν ε, τον αγώνα τους κατά των ε, σεξουαλικών ε, εγκλημάτων βάσει του άρθρου 208 παράγραφος 1. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για μια μάστιγα που πλήττει κυρίως στις υπονάπτυξη χώρες. Στο Κονγκό, για παράδειγμα, και ξέρουμε και έχουμε στο μυαλό μας όλη την μαρτυρία του γιατρού Μουκβέκητς, γυναικολόγου, που ίδρυσε μια ειδική κλινική για γυναίκες που είναι θύματα βιασμών στο νότιο Κίβου και ο οποίος ήρθε και μας προσέφερε τη μαρτυρία του αυτή εδώ το Μάιο. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να αναγνωρίζονται ε, τα θύματα και να διώκονται οι θύτες. Είναι μεγάλη πολιτική μας προτερότητα αυτό. Επίσης θα ήθελα να καθίσουμε και να σκεφτούμε λίγο την ε, ιδέα για να θεσμοθετηθεί η έννοια του εγκληματικού, ε, μάλλον του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Γιατί και αυτά είναι εγκλήματα πολύ συχνά σε βάρος αυτόχθονων πληθυσμών, οι οποίοι εξαφανίζονται και αυτοί και τα μέρη τους αν τίποτα δεν γίνει. Να λοιπόν κάποιες ιδέες που έχω και από εκεί και πέρα ε, ό,τι τροποποίησεις θέλετε να επιφέρουμε στο κείμενο παρακαλώ στη διάθεσή σας να μου το πείτε. Δεν βλέπω να θέλει το λόγο. Α, ο κύριο Γκέρεν. Παρακαλώ κύριε Γκέρεν. Ευχαριστώ. Καταρχήν συμφωνώ με όσα μας είπατε και τις ε, προτάσεις σας. Τις στηρίζω. Όμως θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο περισσότερο την πτυχή που συνδέει την ε, αναπτυξιακή μας πολιτική με τα οικονομικά συμφέροντα. Εδώ νομίζω ότι χρησιμοποίησατε μια γλώσσα κάπως ομή. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, με ποιο τρόπο. Τι στάση πρέπει να υιοθετούμε, άπαξ και θέλουμε να ε, βαρύνει η ζυγαριά προς την σωστή πλευρά και όχι τη λάθος. Πρέπει να δούμε κάθε φορά ποιος είναι ο συσχετισμός δυνάμεων Αντί λοιπόν να λέμε ότι δεν θα λαμβάνουμε υπόψη τα οικονομικά συμφέροντα, εγώ θα προτιμούσα να μιλήσουμε για μια πολιτική μικρών βημάτων. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνηθίζουμε να λέμε ότι ο διαρθρωμένος διάλογος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κίνα δεν φέρει αποτελέσματα. Δεν είναι αλήθεια, γιατί αυτός ο διάλογος έχει κάνει την Κίνα να αλλάξει στάση δεδομένου ότι έχει δεχτεί διάφορε νομολογίε. που σημαίνει ότι ορισμένοι ελευθερώθηκαν που ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο και έχουν δικαίωμα σε νέα δίκη. Δεν λέω ε, από τις απαιτήσει μας, απέχουμε βέβαια έτη φωτός. Παρόλα αυτά είναι μία πρόοδος. Γι' αυτό θα έλεγα, αντί να αναφερόμαστε σε αυτό το ψήφισμα, σε αυτό που είπατε εσείς. Εγώ θα ήθελα να το ζυγίσουμε καλύτερα και να προωθήσουμε την πολιτική αυτή των μικρών βημάτων. Αν το πλαίσιο έχει ετεθεί, με μικρά βήματα μπορούμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Να συγκλίνουμε δηλαδή προς το τελικό μας στόχο με μικρά βήματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει μήπως το λόγο. Έχει κάτι να πει σχετικά με την γνωμοδότηση αυτή. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώ. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τώρα ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι ένα σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε όλοι να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ κύριε Γκέρενς. Κύριε Πρόεδρε, έχω μία πρόταση συγκεκριμένη για τη συνέχεια των εργασιών μας. Νομίζω ότι προχωράμε γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε ολοκληρώσει πριν από την ώρα των ψηφοφοριών, έτσι όπως έχει προβλεφθεί. Μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε νωρίτερα την ψηφοφορία και νωρίτερα τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών ώστε να είμαστε όλοι εδώ και να μπορέσουμε έτσι να τελειώσουμε και νωρίτερα. Πρόεδρος, μου φαίνεται δύσκολο να αλλάξει η ώρα της ψηφοφορίας, γιατί υπάρχουν ευρωβουλευτές που προβλέπουν να φτάσουν την ώρα που έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία. Μήπως τότε τους συντονιστές να τους ξεκινήσουμε νωρίτερα, να σταματήσουμε για τη ψηφοφορία που θα πάρει λίγο έτσι κι αλλιώς και μετά να συνεχίσουμε με τους συντονιστές. Τι θα λέγατε. Είναι περίπλοκο αυτό που ζητάτε, γιατί οι συνεδρίες των συντονιστών είναι και κλεισμένο το θυρών. Για τα γεννόσιμα φάρμακα έχουμε ακόμα ένα σημαντικό θέμα. Ίσως το σημείο 12β να το δούμε τώρα που είναι τα γεννόσιμα φάρμακα. Συμφωνείτε? Καλώς, ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 12α. On était Συγγνώμη, αλλά δεν είναι εδώ ο αρμόδιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξετάσουμε τώρα το σημείο αυτό 12α. συνεπω δεν μπορούμε. Ο κυριο Μαρτίνες. Να ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη. Ας προχωρήσουμε με το επόμενο σημείο που είναι το σημείο 10. Αν έχουμε χρόνο τότε στη διάθεσή μας, μετά το σημείο 10 δηλαδή, τότε βλέπουμε. Δεν ξέρω πόσο θα μας πάρει αυτό το σημείο. Πέντε λεπτά, μισή ώρα, δεν ξέρω. Αν μετά το σημείο 10 παρόλα αυτά μένει χρόνος μέχρι τις προφορίες, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το 12α. Στο κάτω-κάτω έτσι μπορούμε και να ειδοποιήσουμε τον αρμόδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει λίγο νωρίτερα. Αλλά ας κάνουμε πρώτα το σημείο 10. Αυτό είναι στη σειρά. Πρόεδρος, ναι, ναι, σωστά. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. sur Περνάμε στο σημείο 10 λοιπόν, εργασίε τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση ίση εκπροσώπηση ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα κλασικό θέμα γιατί είναι μια έκθεση που κάθε χρόνο εξετάζουμε και ψηφίζουμε και που έχει να κάνει με τι εργασίε τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση ίση εκπροσώπηση τη προηγούμενη χρονιά. Πέρυσι εγώ είχα υποβάλει την έκθεση αυτή για το 2009. Τώρα για το 2010 η συγγετής μας είναι ο κύριος Κάσμαρεκ. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κύριε Κάσμαρεκ. Αλλά προηγουμένως να σας γνωστοποιήσω ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στην γαλλική ε, μετάφραση γιατί εκεί που μιλάνε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωση στις παραγράφους 2 και 14 δηλαδή του σημείου αυτού. Εντάξει, θα διορθωθεί. Κύριε Κάσμαρεκ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια έκθεση, όπως είπατε και εσείς, που επαναλαμβάνεται. Την κάναμε και πέρσι και την κάνουμε και φέτος. βασιζόμαστε στις αρχές της Συμφωνία του Κοτονού. Η κοινοβουλευτική αυτή συνέλευση ίση εκπροσώπηση έχει πολύ μεγάλη σημασία και για μας και για τους συναδέρφους μας από τις χώρες ΑΚΕ. Το 2010 είχαμε δύο ολομέλειες, στην Τενερίφη και στην Κινσάσα, δηλαδή σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν. Και στι Εχέλε έγινε μια περιφερειακή συνεδρίαση. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης εκπροσώπηση επίση συνεδρίασε και στη Μαδαγασκάρη και στην Αϊτή πληροφοριακά και έγινε και μία αποστολή παρατήρηση των εκλογών στον Μπουρούντι. Αυτό που, είναι, ήταν σημαντικό το 2010 ήταν ότι άλλαξε η δομή των Ολομελιών. Βγάλαμε μία μέρα από τις Ολομέλειες, οπότε ε, μειώθηκε το κόστος της οργάνωσης των κοινοβουλευτικών αυτών συνόδων, κάτι το οποίο σε σχέση βέβαια με την κρίση στην οποία αναφερόμαστε συνέχεια. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και νομίζω ότι το καταφέρνουμε, αν και βέβαια η οικονομία δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να δούμε πώς θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Άλλαξε επίσης και ο κανονισμός των συνεδριάσεων. Έτσι, η ομάδα εργασίας του προεδρίου αλλάζει κάπως. Το θέμα είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στις εργασίες μας στην κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης και οι εργασίες μας εκεί να είναι πιο καρποφόρες. Στην Κιντσάσα δεν υπήρξε κανένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτό ήταν κάτι το οποίο λείψε τους παρόντες εκεί. Τόσοι Ευρωπαίοι όσο και η πλευρά των ΑΚΕ το σχολίασαν πολύ, τη σχολίασαν πολύ την απουσία αυτή. Και λυπούμεθα γι' αυτό. Η αιτιολόγηση ήταν ότι υπήρχε γενίαση κάποιων νέων υπηρεσιών κλπ. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί όμως αυτό ποτέ στη Βουδαπέστη. Για παράδειγμα. Και ελπίζουμε ότι τόσο εμείς οι Ευρωπαίοι όσο και οι χώρες εκεί από την πλευρά τους ότι καταλαβαίνετε πως θέλουμε να είναι πάντα παρόν το Συμβούλιο και μάλιστα σε όσο γίνεται υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης πιστεύω ότι ενισχύει το ρόλο των κοινοβουλίων των χωρών ΑΚΕ με ε, δραστηριότητες ε, ελέγχου, εποπτείας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για μας και για εκείνους. Και με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε ότι είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στη Βαρσοβία το Δεκέμβριο, στη διάσκεψη κορυφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και τη Γραμματεία και κυρίως τον Φρανσίσκο για την βοήθεια που μας προσέφερε ετοιμάζοντας την έκθεση αυτή. Δεν ήταν και εύκολο. Ευχαριστώ πολύ, Φράνσις, για τη δουλειά σου. Επίσης, ό,τι τροπολογίες θέλετε να συμπεριλάβουμε, σχόλια κτλ. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Μαρτίνες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το έργο του κυρίου Κασμάρεκ, για την έκθεσή του δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι ο φίλος Κασμάρεκ είναι ένας από τους πιο τακτικούς πιο μόνιμους και πιο ενθουσιώδης για το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ή της Εκπροσώπησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ενθουσιασμός του αυτός, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πάντα. Βλέπετε, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε στις συνεδριάσεις αυτές ή για να γίνει η πραγματικότητα, δηλαδή η συμμετοχή από πλευρά της Ευρώπης πολύ συχνά λείπουν ορισμένοι αντιπρόσωποι από όλες τις ομάδες και τελευταία στιγμή αναγκαζόμαστε να γεμίσουμε τα κενά από άλλους ευρωβουλευτές που δεν είναι μόνιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς ε, να γνωρίζουν σε βάθος τα διάφορα θέματα. Οι συνομιλητές μας από πλευράς των χωρών ΝΑΚΕ παρακολουθούν το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και είναι πάντα παρόντες. Στις Βρυξέλλες επίσης οδηγηθήκαμε μερικές φορές να μπούμε σε αίθουσα κοινή περίπου. Οι συνάδελφοί μας από τις αφρικανικές χώρες, Καρυβική κτλ. ήταν παρόντες, ενώ οι συνάδελφοί μας απο Ευρωπαϊκή Πλευρά, πλευράς, εκτός από εξαιρέσει τρει, τέσσερι οι υπόλοιποι να λείπουν. Οι άντε ερχόντουσαν στην αρχή και σιγά σιγά φεύγανε. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνοι οι οποίοι ορίζονται από τις ομάδες τους, τις πολιτικές τους ομάδες, ως μέλη τη κοινοβουλευτική αυτής συνέλευσης πρέπει να καταλαβαίνουν ότι έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις εργασίες τη. Δυστυχώ δεν συμβαίνει αυτό μέχρι τώρα. Τώρα κατά τα άλλα η έκθεση αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ και προσφέρει ένα δημοκρατικό πλαίσιο και ανοιχτό πλαίσιο προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο στο διάλογο για θέματα που έχουν να κάνουν με διαπραγματεύσεις για οικονομικές συμφωνίες, για την οικονομική κρίση, κλιματικές αλλαγές ή ακόμα και για την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική ή στη αλλού. Είναι θέματα που σίγουρα έχουν μεγάλη σημασία και που αναμφίβολα αξίζουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τη δικιά μας την πλευρά. Όπως είπε και ο Φίλιπ Κασμάρεκ, οι αλλαγές που, που έλαβαν χώρα στην οργάνωση των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ή εκπροσώπησης, οι αλλαγές αυτές λοιπόν σίγουρα είναι σημαντικές ο κόσμος πολλέ φορέ τον ακούει αλλαγέ, Νομίζω ότι γίνονται τεράστιες αλλαγέ κοσμοστορική σημασίας. Όχι, όχι καθόλου. Πρόκειται για μικρές αλλαγέ, οι οποίες όμως βοηθούν στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα όσον αφορά την οργάνωση των ε, πολιτικών οικογενειών ή των ιδεολογικών οικογενειών. Μέχρι τώρα στην Ευρώπη ξέραμε τις πολιτικές ομάδες. Αυτό γνωρίζουμε εμείς στη δικιά μας την Ήπειρο. Όμως στην αφρικανική πλευρά αυτό το πράγμα λειτουργεί διαφορετικά. Περιφερειακά συγκεντρώνονται οι οικογένειες. Οι συνεδριάσεις των πολιτικών οικογενειών έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία. και δεν μιλάνε για πολιτικές ομάδες. Και μένα μου έκανε εντύπωση που διαπίστωσα πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή τους. Δεν είναι όπως παλιά που εμείς οργανώναμε ένα δείπνο και τους καλούσαμε, ερχόντουσαν να φάνε πολύ ωραίο, όχι τώρα έρχονται, να συζητήσουν Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι προσπαθούν να συμβρίσκονται με εκείνους με τους οποίους θεωρούν ότι έχουν περισσότερα κοινά σημεία. Μέσα στις χώρες ΑΚΕ πρέπει να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για τα πράγματα τα οποία προηγουμένως είχαν συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών οικογενειών. Κάτι άλλο σημαντικό, στο οποίο αναφέρεται στην έκθεσή του Φιλίπ Κασμάρεκ, είναι το πόσο ικανοποιητικές αποδείχτηκαν οι περιφερειακές διασκέψεις. Πολύ πιο ενδιαφέρουσες, ακόμα και από τις ολομέλειες. Οι περιφερειακές αυτές διασκέψεις είναι περιορισμένες, πολύ περιορισμένες στον αριθμό. Συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος από κάθε μία από τις χώρες Αφρικής, Καραβικής, ε, Ειρηνικού και αντίστοιχος αριθμός από εμά. Είναι συνεδριάσεις δηλαδή όπου μπορεί να είναι 8-10 αντιπρόσωποι από τους εταίρους μας και άλλοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο συζητήσεων, επαφών αλλά και παρουσίας από πλευρά της Ευρώπης εκεί, το επίπεδο λοιπόν συμμετοχής είναι πολύ πιο σημαντικό. Γι' αυτό και το λέω και επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή, η παρουσία των Ευρωπαίων στις διασκέψεις αυτές είναι πάρα πολύ καλή και συμμετέχουν εκεί ευρωβουλευτές άντρες και γυναίκες και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερο οι γυναίκες παρούσες από ότι οι άντρες συνάδελφοι. Το λέω. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι μια μικρή σύνθεση οι διασκέψεις αυτές, αλλά αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε την ε, παρουσία και τη συμμετοχή των γυναικών εκεί. Τέλος, ένα τελευταίο σχόλιο που μπορεί να μην είναι political correct για να το βάλουμε στην έκθεση, αλλά εγώ το λέω παρόλα αυτά. Ο συντονιστής από πλευρά των σοσιαλιστών στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αυτοκανοποίησή μας. Τι να λέμε, είμαστε εδώ, ο Φιλίπ έκανε την έκθεσή του, τη βλέπει η Επιτροπή μας, η Ολομέλεια την εγκρίνει και πάμε παρακάτω. Μα δεν είναι δυνατόν οι συνάδελφοι που 99% των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενημερώνονται ούτε τους απασχολούν τα θέματα τα οποία εδώ συζητάμε. Η συνθήκη Κοτονού δεν είναι μια οποιαδήποτε συνθήκη, είναι συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 78 χώρες οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης θα είναι και είναι ήδη εταίροι μας και όσον αφορά την πολιτική, όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο και την πολιτική. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στέλνει μια αντιπροσωπεία που μεταξύ μας να τα λέμε, να τα βρίσκουμε, ενώ οι περισσότεροι από τους συναδέρφους μας δεν έχουν την παραμικρή περιέργεια, ούτε την παραμικρή ανησυχία και ούτε την παραμικρή ενημέρωση για το τι συζητάμε. Είναι όπως με τη Λατινική Αμερική, με τη Μεσόγειο, αλλά επιπλέον εδώ μιλάμε για 78 χώρες του νοτίου ημισφαιρίου που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις σχέσεις βορρανότου οι περισσότεροι συνάδελφοί μας δεν παρακολουθούν καθόλου ούτε τις εκθέσεις ούτε τίποτα. Είναι ένα θέμα που περνά παρατήρητο εντελώς στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Δεν ξέρω πως θα πρέπει από τις πολιτικές ομάδες να γίνει μια προσπάθεια εμείς να ενημερώνουμε τους συναδέρφους και να μην ε, νιώθουμε ικανοποιημένοι επειδή οι εκθέσεις μας περνάνε ε, με ομοφωνία Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι εγώ παρουσίασα την πρώτη. Ε, πάντα ομόφωνα εγκρίνονται οι εκθέσει αυτέ. Γιατί? Όχι τόσο γιατί ο κόσμο ενδιαφέρεται και όντω συμφωνεί, αλλά γιατί πολιτικά είναι ορθό να εγκρίνει κανεί τέτοιε εκθέσει. Χωρί όμω να ξέρουν περί τίνο πρόκειται. Και μάλιστα έτσι στην έκθεση αυτή εγκρίνουμε πράγματα που μετά έρχονται σε αντίθεση με άλλα πράγματα που λέει για παράδειγμα μια έκθεση της Επιτροπής ε, Εμπορίου ή δεν ξέρω εγώ τι. Παρόλο που ομόφωνα έχουμε γκρίνει αυτή την έκθεση. Για παράδειγμα ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη πρέπει να έχει κοινοτικό χαρακτήρα. Ωραία. Το ψηφίζουμε, περνάει σε τέτοιες ε, δεύτερες κατηγορίες ψηφοφορίας κατά κάποιο τρόπο και μετά φτάνουμε και αντιφάσκουμε αυτό που έχουμε ψηφίσει. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την υπομονή σας και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Φιλίπ ε, Κασμαρέκη για την ε, έκθεση που μας παρουσίασε και συζητάμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρτίνες. Το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γκοέρενς, θέλετε κάτι να πείτε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο φίλος μου Άγγελ, απλώς θέλω να κάνω μία ερώτηση στον εισηγητή, διότι τελευταίως δεν έχω παρακολουθήσει από κοντά τις σχέσεις και τις εργασίες με τις χώρες ΑΚΕ και αναφέρουμε στις μη ευρωπαϊκές χώρες ΑΚΕ. Έχουμε μιλήσει για τον προϋπολογισμό του θέματος αυτού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 ε, δεν ε, ξέρω αν ε, έχει κοστολογηθεί το θέμα του Ταμείου Ανάπτυξης διότι πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ιδίως όσον αφορά την συνειδιοκτησία του Ταμείου μεταξύ χωρών και, και Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, μπορεί να ε, έχει, έχει εξεταστεί τι γίνεται στο τομέα αυτό με τις χώρες και στο μέλλον ε, εφόσον θα γίνει αυτή η συμπερίληψη στον προϋπολογισμό θα προχωρήσουμε έτσι κάποιος θα πρέπει να το κοιτάξει για να γνωρίζουμε αν υπάρχει απλώς μία απλή διαδικασία ECI οπότε θα χαθεί η επιρροή μας σε αυτές τις χώρες και πιστεύω ότι στο θέμα της συμμετοχικής ε, ε, ε, συμμετοχής θα έπρεπε να δούμε πώς θα ρυθμιστεί το θέμα αυτό και προτού καθοριστούν ε, τελεσίδικα οι προοπτικές για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο να το έχουμε υπόψη μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο μέσω της κυρίας Κάτριν Μέτιεν Πίνιγκεν. Έχουμε ορισμένα σχόλια σχετικά με την έκθεση σε γενικές γραμμές ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα σχόλια που έχουν γίνει ε, διότι Προσπαθούμε να υπάρχει πλήρη έκφραση των δημοκρατικών αρχών και κοινοβουλευτικών απόψεων αλλά δεν συμφωνούμε επί της ουσίας διότι συνεργαζόμαστε όσον αφορά το θέμα αυτό με τα εθνικά κοινοβούλια έχουμε ορισμένες, ορισμένους πόρους οι οποίοι ε, χρησιμεύουν στην προώθηση ε, της ε, συμμετοχικής κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και προσπαθούμε όλα τα στοιχεία να μεταδίδονται μέσω της γραμματείας του GPA όσον αφορά την οικονομική συνεργασία έχουμε κοινά εποπτικά, κοινούς εποπτικούς οργανισμούς, ιδίως ε, στην Καρεβική, για να αξιολογούμε τις επιπτώσεις των δράσεων αυτών στην περιοχή αυτή. Εκεί που έχουμε προβλήματα είναι η διατύπωση ή στο σχέδιο εκθέσεως γιατί ζητείται από την Επιτροπή να εγγυηθεί νομικά την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η Συμφωνία του Κοτονού που συνδέει τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις χώρες ΑΚΕ ε, λέγεται ε, ότι η ομόλογή μας είναι οι χώρες ΑΚΕ και όχι τα κοινοβούλια τους. Νομίζω λοιπόν ότι ο όρος όσο υπερβαίνει τις ε, συμβατικές μας υποχρεώσεις και το, τη θεσμική ουσία του θέματος. Οπότε θέλω να αναφερθώ εις ε, το άλλο θέμα που θίγει, δηλαδή το ότι πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται σωστά η Συμφωνία του Κοτονού που δεν παρουσιάζει βασικά θέματα αλλά στο, στο πνεύμα αυτής της ε, συμφωνίας υπάρχουν ορισμένες φορές προβλήματα και ε, θα επανέλθουμε σε εσά όταν θα έχει προσαρμοστεί η Συμφωνία του Κοτονού στη Συμφωνία της Λισαβόνας. Ε, ο κύριε Κασμάρε, και έχετε το λόγο για να κλείσετε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και τις προτάσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρτίνες ότι ένα από τα προβλήματά μας ιδίως όσον αφορά τις ε, συνεδριάσεις με τους ομολόγους μας είναι η ανεπαρκής συμμετοχή των ε, ευρωβουλευτών και στις συνεδριάσεις οι οποίες γίνονται εις ε, τον οίκο των χωρών και στις Βρυξέλλες είτε εδώ. Δεν μπορούμε βέβαια να εγγυηθούμε αυτή την παρουσία ακόμη και αν ε, έχουμε εισάγει ε, την ε, ε, πρόβλεψη ενός ε, μονίμου πληρωματικού μέλους του Προεδρείου πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την συμμετοχή διότι αν θέλουμε όντως να θεωρήσουμε τις συνεργασίες αυτές σοβαρά θα πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι και να το εκφράζουμε την παρουσία μας. Είναι προφανές. Ε, συμφωνώ επίσης ότι η συμφωνία του Κοτονού πρέπει να παρουσιάζεται καλύτερα στις ε, συζητήσεις μας διότι η αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας απαιτεί τη την συνένεση όλων των κρατών μελών οπότε θα πρέπει όλοι να δεσμευτούμε και να ενδιαφερθούμε από το θέμα αυτό και όλοι οι ευρωβουλευτές θα πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν ποια είναι η ουσία των θεμάτων που μας απασχολούν στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες και ε, τώρα όσον αφορά την ε, περίληψη στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού τα. Ταμείου Αναπτύξεως με τις χώρες ε, ΑΚΕ είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στις συνεδριάσεις και οι χώρες αυτές θεωρούν ότι η οργάνωσή μας δεν ε, είναι η ε, κατάλληλη δηλαδή θα έπρεπε οι δαπάνες να λαμβάνουν υπόψη περισσότερο τις προτάσεις των ομολόγων μας. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν αυτές οι συνεργασίες θα ήταν πιο ουσιαστικές ουσιαστικές για να μπορούμε να ε, προσαρμοστούμε περισσότερο στις χώρες ΑΚΕ. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υπάρχει καλύτερη συμμετοχή των χωρών οι οποίοι ε, υποφελούνται από αυτή τη συνεργασία ε, είναι κάτι που θα πρέπει να καθοριστεί. Αλλά εάν εμπλέκονται τα κοινοβούλια τότε και οι ομόλογοι μας και εμείς ε, μπορούμε να αξιολογήσουμε εάν ε, είναι η σωστή οδός. Το 2010 δεν είχαμε πολλά προβλήματα και υπήρχε μία σαφή στάση να ενισχύσουμε τον ρόλο των κοινοβουλίων και βεβαίως η Συμφωνία του Κοτονού έχει κυρωθεί από τα κράτη, από ολόκληρες χώρες αλλά από τη μία πλευρά είμαστε ικανοποιημένοι να βλέπουμε όλο και περισσότερους ευρωβουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν ε, ε, όλο και περισσότερους βουλευτές με συγχωρείτε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αλλά δεν μπορούν να έρθουν οι βουλευτές μπορούν να αντικατασταθούν με τους ε, πρέσβεις αποτελεσματικά και αντιλαμβάνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υποχρεώσει τις χώρες ΑΚΕ να κάνουν κάτι αλλά εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο από κοινού Κοινοβουλίου τονίσουν ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες να αναβαθμιστούν τα κοινοβούλια. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε από κοινού. Είμαστε ρεαλιστές και γι' αυτό συμφωνούμε οι πρέσβεις να συμμετέχουν στις ε, ε, συνεδριάσεις της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης ή στις εκπροσώπησης. Λαμβανόμαστε ότι μειών αυξάνονται οι πρέσβεις και αυξάνονται οι βουλευτές. Αλλά οι βουλευτές βεβαίως θέλουν ο ρόλος των κοινοβουλίων και από τις δύο πλευρές να αναβαθμιστεί. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε ε, για τις ε, τροπολογίες ε, χρόνο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 22 Σεπτεμβρίου. Έχουμε εδώ μία μία ε, αντιπροσωπεία από συναδέλφους από τον Μπουρούμπι ε, με εκπροσώπους ε, του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας της χώρας αυτή και βρίσκονται εδώ διότι υπάρχει μία έρευνα η οποία καταρτίζεται από το Γραφείο Κοινοβουλευτικών Μελετών και τους καλωσορίζουμε εις αυτήν τη συνεδρίαση. επαναλαμβάνει ε, ένα καλωσόρισμα η πρόεδρος στη γλώσσα του Μπουρούντι υποθέτω. Έχουμε ακόμη πέντε λεπτά μέχρι τις ψηφοφορίες και ξεκινάμε με το θέμα 12β δηλαδή ανταλλαγές απόψεως ε, με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα γενώσιμα φάρμακα και στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ινδίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση ε, του AIDS και έχουμε λάβει επί του θέματος ε, μη ε, ε, αίτηση από την Επιτροπή Αναφορών διότι υπάρχει ο φόβος ότι η μελλοντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα εμποδιστεί να υπάρχει αποστολή των γενοσύμων αυτών φαρμάτων προς υποανάπτυξης χώρες όπως η, ε, το, η Βραζιλία και άλλες. Έχουμε λοιπόν ε, διάφορους εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι θα μας καθησυχάσουν και εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας αποδείξουν ή θα μας πείσουν ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει αυτή η εξέλιξη να υπάρχει μία πρόσβαση στην, ε, στα γενώσιμα φράρμακα. Δίνω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Γέντσεν, ο οποίος έχει το λόγο για 8 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Επιβεβαιώνω εκ μέρους της Κομισιόν ότι πετύχαμε έναν φιλόδοξο στόχο στο FTA με την Ινδία. Παραμένει μάλλον αυτό σημαντικό στόχος όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, ταυτόχρονα, ξέρουμε ότι η Ινδία είναι, παίζει σημαντικό ρόλο ως πηγή γενοσύμων φαρμάκων για άλλε αναπτυσσόμενε χώρες. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας στις διαπραγματεύσεις. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις επιδεικνύουμε ευελιξία Λαμβάνω υπόψη τη ιδιομορφία του νομικού συστήματο στην Ινδία και το ρόλο τον οποίο παίζει η Ινδία στο μέτωπο αυτό. Και γι' αυτό κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για το FTA και ρητή μνήμα στην δήλωση της Ντόχα για τη Συμφωνία TRIPS για τη δημόσια υγεία έτσι ώστε οι ευελιξίες αυτές που εξασφαλίστηκαν μέσω της συμφωνίας DRIPS, ιδιαίτερα όσον αφορά τα, τις για τα φάρμακα, να μην περιορίζονται από τη συμφωνία FTA, όταν θα έχει ολοκληρωθεί βέβαια. Επίσης, προτείναμε στους Ινδούς μια διάταξη που ορίζει ότι στη συμφωνία τίποτε δεν θα ερμηνευθεί ως περιοριστικό της δυνατότητας πρόσβαση στα φάρμακα από όλους τους εταίρους και θα αναφερθώ τώρα στα τρία κύρια σημεία που αναφέρονται στην αναφορά. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για το πρώτο σημείο προστασία πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων. Με βάση την ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται αυτό, αποκλειστική χρήση των πληροφοριών αυτών. Γίνεται συζήτηση στην Ινδία σχετικά με την αποκλειστική χρήση αυτών των πληροφοριών και θα πρέπει να εισαχθεί ή όχι, αλλά επειδή το θέμα αυτό παραμένει ακόμα ασαφές, κατά πάσα πιθανότητα η Ινδία δεν θα έχει εισάγει ένα σύστημα όταν θα έχουν ολοκληρωθεί η διαπραγματεύση για το ΕΦΤΕ. Η Κομισιόν επιμένει ότι το λέμε αυτό και στο site, στην ιστοσελίδα μα και απαντώντα σε ερωτήσει του Ευρωκοινοβουλίου, εμεί επαναλαμβάνω λέμε ότι δεν θα ζητήσουμε από την Ινδία να εισάγει διατάξει για την αποκλειστική χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων στο FTA. Πρόσφατα δώσαμε απάντηση μια γραπτή ερώτηση 002-2442-2011 και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Ο Επίτροπος έγραψε και στους ευρωβουλευτές και στο προς το κοινό γενικότερα και υπάρχουν πολλές απαντήσεις στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Δεν το ζητάμε αυτό από τους Ινδούς. Ίσως δημιουργήθηκε σύγχυση λόγω του ότι υπάρχει ένα ερώτημα η ειδική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, όχι αποκλειστική χρήση, προστασία των προσωπικών δεδομένων, αν συμφωνεί με το 39.2 άρθρο του TRIPS. Οι Ινδοί έχουν κάνει εκθέσεις και τα συζητάνε. Αν θα υπάρξει συμφωνία με την Ινδία, η Ινδία επιβεβαιώνει ότι δεσμεύεται να εφαρμόσει πλήρως το TRIPS. Αυτά για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τώρα, η επέκταση της ε, ε διάρκειας των ευρεσιτεχνιών. Ούτε και αυτό είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Το τελευταίο χρόνο, κατά επανάληψη κομισιών, το έχει πει και προς το Κοινοβούλιο με γραπτές ερωτήσεις. Δεν ζητάμε και δεν θα υπάρχει διάταξη στο FTA η Ινδία να προβλέπει αυτή την επέκταση του όρου χρήσης ευρεσιτεχνιών. Και τέλος, για τα μέτρα για τα σύνορα. Δεν προβλέπεται τίποτα στη διαπραγματευτική θέση να ζητήσουμε δηλαδή από την κυβέρνηση της Ινδίας τα μέτρα αυτά των συνόρων να τα ευθυγραμμίσει με αυτό που ισχύει για μας όσον αφορά τα, τους ε, τελωνιακές ρυθμίσεις. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ινδίας και Βραζιλίας και ζητήθηκε να φύγει μια αιτιολογική σκέψη που θα μπορούσε να ερμηνευθεί έτσι ώστε να, να οδηγήσει σε κατάσχεση γενοσύμων φαρμάκων transit ως προς την Ένωση. Θα φροντίσουμε το κείμενο να συνταχθεί με τρόπο ώστε να υπάρχει, να εξασφαλιστεί μάλλον η συνεχής ροή των γενοσύμων φαρμάκων και οι διατάξεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελέσουν αντικείμετρο στην αφορά τον ανταγωνισμό για τα γενώσιμα φάρμακα ή την εξαγωγή γενοσίμων φαρμάκων σε λοιπές αναπτυσσόμενες χώρες. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της Κομισιόν. Η Κομισιόν αρχικά σκόπευε να βάλει την αποκλειστική χρήση των ευρεσιτεχνιών και την επέκταση των ευρεσιτεχνιών να τα βάλει στο κείμενο και επίση το κοινοβουλίο εξασφάλισε ότι δεν θα είναι στο τελικό κείμενο. Η κατάσταση σχετικά με τα γενώσιμα δεν είναι τέλεια. Τα TRIPS ήδη αύξησαν τις τιμές για τα γενώσιμα, αρκετά μάλιστα, και από ό,τι ξέρω Στη συμφωνία με την Ινδία θα αναφέρεται ότι από τη στιγμή που η Ινδία θα εισάγει την αποκλειστικότητα των προσωπικών δεδομένων, αυτό θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Είπατε ότι τίποτε δεν θα παραβλάψει την παραγωγή και την εξαγωγή ουσιωδών φαρμάκων. Θα ήθελα να μας δώσετε ένα ορισμό. Τι εννοείται όταν λέτε ουσιώδη φάρμακα, essential τι είναι αυτά που σώζουν ζωές, ε, φάρμακα, τι είναι, πόσο το ορίζεται το ουσιώδες φάρμακο. Ακούμε πολλά, πολλές φήμες κυκλοφορούν, τίποτα σαφές δεν υπάρχει στο τραπέζι ακόμα. Καλό θα είναι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να μας δώσει στην Επιτροπή μας τα διαπραγματευτικά έγγραφα, τα κείμενα να δούμε αν έχετε δίκιο ή όχι, αν χρειάζεται να διορθώσουμε ή όχι τη θέση μας. Πώς να το κάνουμε αυτό, αν κυκλοφορούν μόνο ασαφείς φήμες από εδώ και από εκεί. Επίσης θα έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη αν διαπιστώσουμε ότι και η άλλη γενική διεύθυνση παίρνει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Η γενική διεύθυνση DEF θα πρέπει και αυτή να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις αυτές έτσι ώστε να δοθεί μια διαφορετική προοπτική διότι η Ινδία είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό φτωχών. Τέλος, τι θα κάνετε προκειμένου να εισηχθεί μια αξιολόγηση επίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί το προτείναμε και η Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι θα κάνει μια αξιολόγηση επίπτωση σχετικά αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τα γενώσιμα φάρμακα και με άλλα θέματα. Γιατί πέραν του πολύπλοκου αυτού θέματος των γενοσύμων, το FDA προτείνει ή αποτελεί κίνδυνο και για άλλα θέματα όπως η απασχόληση, η διακυβέρνηση. Θα ήθελα να μας πείτε αυτή η αξιολόγηση επίπτωση αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που μας υποσχεθήκατε πότε θα την έχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Γέσεν, δύο λεπτά σας παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Το σημειώνω και θα το μεταβιβάσω στους συναδέλφους μου για την εμπλοκή της Επιτροπής σας. Εμείς ως Γενική Διεύθυνση Εμπορίου σεβόμαστε τις διατάξεις της δια... συμφωνία, συμφωνίας, διοργανικής συμφωνίας και ό,τι έγγραφα έχουμε, ό,τι προβλέπει η συμφωνία, σας τα δίνουμε. Αν είμαστε φιλόδοξοι ή όχι. Έχουν περίπου 6-7 επιστολές ήδη για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν δημόσια το έχει δηλώσει. Έχουμε γράψει κοινά άρθρα με τον Ινδό Υπουργό Εμπορίου. Το τονίζουμε και το υπογραμμίζουμε το σημείο αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει αμφισημία πια και οι Ινδοί ενδιαφέρονται εξίσου για το θέμα αυτό και περισσότερο μάλιστα από εμά. Συμφωνούμε όμω και σε σχέση με αυτό που ζητάμε. Δεν υπάρχει διαφορά απόψεων. Τι παραπάνω να κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε κι άλλο την κατάσταση. Αποκλειστική χρήση προσωπικών δεδομένων γιατί ισχύει για τα ουσιώδη φάρμακα ή για όλα τα φάρμακα, το θέμα, είπα, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Το έχουμε συμφωνήσει με τους Ινδούς. Οι επέκτες των διατάξεων στο ΕΠΑ ελέγχονται με βάση την τρέχουσα νομοθεσία. Από τη στιγμή που η νομοθεσία δεν έχει αυτή την αποκλειστικότητα στο σύστημά της, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Είμαι νομίζω μέσα στα δύο λεπτά μου και απάντησα. Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε διμερώς τις διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα θα ψηφίσουμε. Σημείο 11 δηλαδή στην ημερήσια διάταξη. Ψηφίζουμε. Α, προηγουμένως πρέπει να σας ρωτήσω. Έχετε τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία μαζί σας. Για ετοιμάστε Θα κάνουμε μια δοκιμή πρώτα για να μετρήσουμε πώς ψηφίζουμε με την ηλεκτρονική κάρτα. Λοιπόν, ψηφίστε παρακαλώ δοκιμαστικά. Ψηφίσατε όλοι. Μια ψήφος λείπει ακόμα. Εντάξει, τώρα ψήφισαν όλοι. Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν και ψηφίζουμε την γνωμοδότηση του κυρίου Γκέρενς όσον αφορά τις αλληλευτικές δυνατότητες στο πράσινο κροτήρι. Ηλεκτρονική ψηφοφορία είπαμε, έτσι. 74 σκάφη επιτρέπεται για 5.000 τόνους. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Συνεπώς, ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Στη συνέχεια έχουμε το σημείο 12, πάντα του κυρίου Γκέρεντς, αυτή τη φορά για τον προπολογισμό. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 5439. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Δύο πρέπει ακόμα να ψηφίσουν. πέρα της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ. 54-38 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. 22 ψήφοι υπέρ. 54-21 τώρα. Ψηφίστε. Α, έχει πέσει. Τροπολογία 54-01. Ψηφίστε. 22 ψήφοι υπέρ. Α, και τρεις αποχές. Και 7 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54-30 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 21 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54-31. 54-32 διορθώνει ο Πρόεδρος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Κύριε Γκέρεν, θέλετε το λόγο. Για να γίνει κάπως πιο εύκολη η δουλειά μας. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε ψηφοφορίες συγκεντρωμένες. Νομίζω ότι συμφωνούν οι περισσότερες πολιτικές ομάδες με τις τροπολογίες που ψηφίζουμε. Οπότε μπορείτε να ρωτάτε τις ομάδες που δεν συμφωνούν με τις τροπολογίες και εκεί όπου υπάρχουν διαφωνίες να ψηφίζουμε χωριστά. Αλλά εκεί που υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων να συγκεντρώνουμε τις ψηφοφορίες και να ψηφίζουμε μια φορά για πολλές μαζί. Πρόεδρος. Τροπολογία 5400. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνονται. 54-04 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. 54-11 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. 54-12. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. δεκατριά ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε υποφορία. Εγκρίνεται. Ίσως τώρα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 5414 μέχρι την 5436, συμπεριλαμβανομένες της 5436. Συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές τις τροπολογίες. Ψηφίστε παρακαλώ. 5414 έως και 5436. Ψηφίσατε όλοι. Πέρες προφορίες. Εγκρίνονται ομόφωνα. Τώρα ψηφίζουμε 5440 Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι οι ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 54-41. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-42 και 54-43 μαζί. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τώρα 54-35. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προτείνω να ψηφίσουμε τώρα την 5423 μέχρι την 5415 συμπεριλαμβανομένης. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο, παρακαλώ. Ψηφίστε. Μία ψήφος περιμένει ακόμα. Περιμένουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας.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 Υπάρχει ένα θέμα στα διάφορα στην ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε όμως ε, διάφορα και μπορώ να σας πω ότι αύριο στις 9 οι συντονιστές θα έχουν μία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κρίστοφ ε, Στανόφσκι υφυπουργό της Πολωνίας ε, και υπεύθυνο για θέματα αναπτύξεως και θα έχουμε επίσης ε, την ακρόαση σχετικά με την παιδεία και την ανάπτυξη από τις 10 ως τις 12 και 30. Η επόμενη συνεδρίαση, τακτική τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα συνέλθει στις Βρυξέλλες τις 22 Σεπτεμβρίου και τώρα θα συνεχίσουμε με την συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν όλα τα άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να αποχωρήσουν από την αίθουσα. και οι συζητήσεις θα μπορέσουν να συνεχιστούν εκτός εθούσης.